μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας του άρθρου 138 του κανονισμού για την έκθεση του κυρίου Σκέρια για το έτος του εθελοντισμού. Ο εισηγητής θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Σκούρια. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις προσπάθειές τους, να ευχαριστήσω όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που εργάστηκαν, όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους εισηγητές που έχουν προσφέρει στην έκθεση αυτή. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο του εθελοντισμού. Εκατό εκατομμύρια Ευρωπαίοι ασχολούνται με, τις, με τους συλλόγους και τις δραστηριότητες αυτές και καθημερινά χωρίς καμία αμοιβή βοηθούν τους συνανθρώπους τους. Λοιπόν, εμείς αυξήσαμε τον προϋπολογισμό, αυξήσαμε τον αριθμό των δραστηριοτήτων, βοηθούμε τους συλλόγους κτλ. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία για την προσπάθεια την οποία κάναμε από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για τον τομέα αυτό που για πολλούς αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της κοινωνίας μας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Has everybody voted? Has everybody voted? The vote is now closed. And that is adopted. Τέλος της ψηφοφορίας γίνεται δεκτό το ψήφισμα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία στην έκθεση Royal για την τεχνική και επιστημονική συνεργασία με την Ουκρανία. Ονομαστική ψηφοφορία ξεκινάμε. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Να παρακαλέσω να διευκρινιστεί ότι και τις δύο φορές ψήφισα ναι, να το σημειώσετε. Ναι, θα το σημειώσουμε, λέει η Πρόεδρος. Το επόμενο θέμα, σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία, έκθεση του κυρίου Ρόιλ, για την διεθνή εταιρική σχέση στον τομέα της αποτελεσματικής ενέργειας και συνεργασίας. Ονομαστική ψηφοφορία ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για τις δύο εκθέσεις. Το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη στρατηγική διεύρυνση για το 2009. Παράγραφος 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τοπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Βεβαίως. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτό. Τροπολογία 12. Ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 11, ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. 11. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην 13. Ποιοι είναι υπέρ της 13. Κατά. Ονομαστική ψηφοφορία από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Όχι. Για μια στιγμή. Ποιοι είναι υπέρ της 4. Ποιοι είναι κατά της 4. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4. Ξεκινάει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ονομαστική. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 14. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Παράγραφος 22. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Παράγραφος 8, ποιοι είναι υπέρ, ε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να υπάρξει έλεγχος για την τροπολογία 8. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία 8. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10. Είναι υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 10. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Η αιτιολογική σκέψη C Χωριστή ψηφοφορία κατά τμήμα. Πρώτο τμήμα, ψήφι κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το ψήφισμα, ο σύνολο, ψήφι κατά, αποχές, δεκτό.